δεν υπάρχει στα εθνικά κοινοβούλια. Πρέπει λοιπόν να επικοινωνήσουμε, να υπάρξει μια διαδικασία επικοινωνία και με τα εθνικά κοινοβούλια. Σα ευχαριστώ κύριε Καράς. Έληξε η συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο για το θέμα αυτό. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Ο κύριος Μπαρνία θα μείνει μαζί μας όλο το βράδυ. Τώρα είμαστε στη δήλωση της Επιτροπής για την επιβολή προστήμων από την Επιτροπή σε υποθέσεις παράβασης των αντιμονοπολιακών κανόνων. Έχετε το λόγο κύριε πίτροπε. Ευχαριστώ, είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι μαζί σας και σήμερα. Εκ μέρους του Ακίμ Αλμούνια που έχει δείπνο εργασίας με την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, εκ μέρους του λοιπόν ήρθα εγώ να σας μιλήσω για το θέμα αυτό προστίμων όταν πρόκειται για παραβάσεις αντιπο, αντιμονοπολιακών κανόνων. Ξέρετε ότι η Επιτροπή καταπολεμάει τέτοιες παραβάσεις εφόσον πλήττουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μέσα στην εσωτερική αγορά και την ενία αγορά. Επιβάλλουμε λοιπόν παραβάσεις, ε, επιβάλλουμε πρόστιμα για τις παραβάσεις που κάνουν επιχειρήσεις που επωφελούνται από την ε, μονοπωλιακή τους θέση. Γίνεται υπολογισμό βέβαια των ε, προστήμων. Πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε κάνει τους πρώτους υπολογισμούς. Ε, μειώνουμε τα πρόστιμα για επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί μας και προσπαθούμε να πετύχουμε μια συμφωνία με τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες ε, δέχονται να συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως. Δεν υποχρόνται να δώσουν πάνω από 10% του τζίρου τους, που αποτελεί όριο για τα πρόστιμα που επιβάλλονται. Τα πρόστιμα είναι το κύριο μέσο πάντως που έχουμε στη διάθεσή μας, χωρίς να αποκλείεται στο μέλλον να επιβάλλουμε άλλες κυρώσεις για τα άτομα, διοικητικές κυρώσεις, μια που πολλά κρατημέλη έχουν ήδη τέτοιε κυρώσει. Εμείς θέλουμε να εξετάσουμε τι νομικέ επιπτώσεις έχει κάτι τέτοιο. Πρέπει τώρα να προτείνουμε ένα επίσημο νομικό πλαίσιο. Είναι το άρθρο 23 του κανονισμού 1 του 2003 του Συμβουλίου που αποτελεί τη νομική βάση των προστήμων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι οι κατευθυντήριε ε, γραμμέ για τον υπολογισμό των προστήμων. Ε, αυτό το 23 βάζει την οροφή όπως σας είπα, σε σχέση με τον τζίρο και οι καθεντήριες γραμμές μιλούν για τον τρόπο εφαρμογής των προστήμων αυτών. Μέσα στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές ε, κυρώσεις που επιβάλλονται. Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα και πρέπει να μελετηθεί για να δούμε εμεί τι αποφασίσουμε. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία έχουν τέτοιε κυρώσει όταν πρόκειται για στρέβλωση του ανταγωνισμού. Βάσει αυτή τη κατάσταση, λοιπόν, εμεί δεν βλέπουμε κανένα λόγο να επιβάλλουμε νέα νομοθεσία στα πρόστιμα αυτά όταν πρόκειται για αντιμονοπολιακούς κανόνε. Τώρα για τι κατευθυντήριε ε, γραμμέ πρέπει να τι δούμε περισσότερο και να σα μιλήσω λίγο για αυτέ πριν ε, φτάσουμε στι κυρώσει. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει μα, η ζημιά που επιβληθεί από τι 10 συνονοήσει που έγιναν ήταν 8 δις ευρώ. Οι μελέτες έδειξαν μάλιστα ότι είχε αυξηθεί το ποσό κατά 10 με 30%. Είναι μια τάση λοιπόν στην οποία πρέπει να αντισταθούμε και άρα πρέπει να φροντίσουμε να εφαρμόζεται αυστηρά κάθε κανόνας για στρέβλωση ανταγωνισμού. Πρέπει να τιμωρούμε κάθε παράνομη συμπεριφορά με σωστό και δίκαιο τρόπο. Τα πρόστιμα είναι υψηλά, αλλά αντικατοπτρίζουν τη ζημιά που γίνεται. Θέλουμε να είναι και αποτρεπτικό μέτρο, ώστε επιχειρήσεις να μην επαναλαμβάνουν τέτοιου είδους ε, μονοπωλιακές ε, συμπεριφορές και όλα αυτά όπως σας είπα βάσει και των κατευθυντηρίων γραμμών του 2006 που κανονίζουν τα πρόστιμα. Τώρα, είμαστε σε κρίση, ναι. Γι' αυτό και εξετάζουμε πάρα πολύ σοβαρά την οικονομική κατάσταση των διαφόρων επιχειρήσεων μερικές φορές όντως δεν μπορούν να πληρώσουν. Οπότε μειώσαμε τα πρόστιμα σε σημαντικό βαθμό για πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις. Πιο, πολύ πρόσφατα πήραμε κάποια απόφαση για είδη υγιεινής, για το χάλιβα. Εφαρμόσαμε εκεί μειώσεις της τάξης 25 με 75%. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν μας εφέρει να αποκλείσουμε από την αγορά τις επιχειρήσεις. Καθ' άλλο. Συχνά οι κανόνες ανταγωνισμού έχουν σαν σκοπό να επιτρέψουν σε νέες επιχειρήσεις να μπουν στην αγορά και να ασκήσουν ε, σωστά και δίκαια τις δραστηριότητές τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Πρώτα και δύο λεπτά, κύριος Λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την Κομισιόν για την ευελιξία που έδειξε. Ο κύριος Μπαρνιέ είπε πως ε, ειδικά στον τομέα των οικοδομών επειδή υπήρχαν ε, κάποια προβλήματα υπήρξε μια ανάλογη αντίδραση της ε, Κομισιόν για να λάβει υπόψη την δεινή οικονομική κατάσταση ορισμένων ε, τέτοιων επιχειρήσεων. Αλλά βεβαίως πρέπει να τεθεί το ερώτημα μήπως το σύστημα της επιβολής ε, των ε, ποινών ε, δεν ανταποκρίνεται πλέον στην νομική βάση. Εγώ τολμώ να πω πως μπορούμε να αμφιβάλλουμε, γιατί βεβαίως ο οργανισμός του 2003 δίνει στην Κομισιόν ένα τόσο ευρύ πεδίο δράσης χωρίς να ορίζει κριτήρια που μπορεί να υποθέσει κανείς πως θα μπορούσε να μην ε, είναι και μη υποχρεωτική απόφαση. Δυστυχώς το Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο μέχρι στιγμής ε, δεν ε, έχει φέρει καμία αντίρρηση. Μπορεί όμως προσεχώς γιατί ξέρετε πως θα τεθεί ενισχύ και η Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα μπορούσε ίσως από εκεί να αμφισβητηθεί αυτή η διαδικασία. Οπότε θα μπορούσε η Κομισιόν είτε να εξετάσει κριτήρια είτε να σκεφτεί άλλο είδος ε, κυρώσεων για να ενισχύσει και να καταστήσει πιο συγκεκριμένη την 1 του 2001 κάτι το οποίο νομίζω είναι απαραίτητο και κάτι το οποίο νομίζω θεωρούν και όλοι οι ειδικοί στον τομέα αυτό στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σάντσες Πρεσέδο τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Μπαρνιέ, το θέμα των προστήμων είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι η αντίδρασή μας σε στραβές συμπεριφορές και πρέπει όντως να είναι αυστηρά και αποτελεσματικά και πρέπει να αποτελούν κίνητρο για να αποφεύγονται παραβάσεις. Όμως τα πρόστιμα πρέπει να είναι και αποτρεπτικά. Αποτρεπτικά για τους παραβάτες, αλλά και γενικά αποτρεπτικά για όλους τους φορείς. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν φέρνει κανένα πλεονέκτημα και κανένα κέρδος η παράβαση των κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βέβαια ένα περιθώριο ελιγμών, μια διακριτική ευχαίρεια, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγονται τα πρόστιμα, γιατί υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν όροι, υπάρχουν κριτήρια, υπάρχει και μια διαδικασία και βέβαια και ένας έλεγχος. Στον ε, κανονισμό αυτόν 1-2003 και σκατζερή γραμμές του 2006, όλα αυτά αποτελούν ένα πλαίσιο που λειτουργεί αρκετά καλά. Όμως το σύστημα επιδέχεται βελτιώσεις. Η εμπειρία μας, η επιχειρηματολογία των εμπειρογνωμόνων, οι ανησυχίες που εκφράζονται από διάφορους φορείς μας οδηγούν να εξετάσουμε το θέμα της διαφάνειας. Μπορούμε επίση να δούμε πάλι τις επιπτώσεις που έχουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιπτώσεις που έχουν τα πρόστιμα αυτά στην απασχόληση να δούμε και την διάρθρωση με προγράμματα και τις αποκλήσεις που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Μπορούμε ίσως να συμπληρώσουμε το θέμα αυτό και με άλλα μέτρα. Να αποφασίσουμε για την ατομική ευθύνη ή να βρούμε άλλα μέτρα για να σταματήσουν αυτές ε, οι μονοπωλιακές συμπεριφορές και να φροντίσουμε για αποζημιώσεις και συλλογικές και ατομικές. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα βλέπουμε συστηματικά. Δεν πρέπει να αφήνουμε αμφιβολίες για το πόσο καλά λειτουργούν οι κανόνες αυτοί. Ευχαριστούμε κυρία Χετβέλτ, έχει τώρα το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προσυπογράφω ε, τα περισσότερα από αυτά που είπαν οι προλήσαντες συνάδελφοι ε, και επίσης ε, και με τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί διαβάζοντας προσεκτικά ε, και ακούγοντας προσεκτικά τα λόγια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, καταλαβαίνω ότι εστερνίζεται ε, τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την καταπολέμηση των ε, ε, μονοπωλιακών ε, κανόνων. Εδώ θέλουμε όχι μόνο επιβολή προστήμων αλλά ένα σύνολο μέτρων που θα αποτρέπει τις ε, ε, στρεβλώσεις του ανταγωνισμού γιατί όπως είπατε και εσείς τελικά ε, αυτό το σύστημα, αυτές οι πρακτικές οδηγούν σε μεγάλη αύξηση τιμών και επομένως αποβαίνουν κακές για τους καταναλωτές. Επομένως ακόμα και αν αλλά βεβαίως να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο και να έχουμε υπερβολικά ψηλά πρόστιμα τα οποία θα γονατίσουν τις επιχειρήσεις και δεν θα μπορέσουν να μείνουν μέσα στον ανταγωνισμό εμείς θέλουμε και μέτρα τα οποία θα καλύπτουν ε, την, ε, ε, την προσωπική ευθύνη, της, την δυνατότητα την δυνατότητα λογοδοσίας ε, κτλ. Ε, βεβαίως θέλουμε να φτάσουμε σε ευρωπαϊκά πρότυπα και θέλουμε να, να μας πει η Επιτροπή πού έχει φτάσει με τις προτάσεις της και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι το θέμα εδώ είναι περίπλοκο γιατί ε, παρότι έχουμε ένα κοινό στόχο να λειτουργήσει καλύτερη αγορά υπάρχουν και οι εθνικές αρχές και οι ευρωπαϊκές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκοζές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια κύριε Επίτροπε είχα θέσει το ερώτημα στον τότε Επίτροπο υπεύθυνο για θέματα ανταγωνισμού. Ε, του είπα λοιπόν έχετε καταλάβει ε, τι χρήσιμότητα έχουν για τους ε, καταναλωτές αυτά τα πρόστιμα ε, και η Επίτροπος μας είχε πει «Μα εγώ πήρα τόσα χρήματα από τα πρόστιμα, αλλά αυτό περίμενα να μου πει, αλλά τελικά εκείνη μου είπε «Όχι, όχι, δεν έχουμε κανένα μετρήσιμο αποτέλεσμα». Θα ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι ο καθορισμός ε, γίνεται βάσει του κύκλου εργασιών του ομίλου, αλλά ε, μια επιχείρηση η οποία ενδεχομένως έχει υποπέσει σε σφάλμα ανταγωνισμού ε, ενδεχομένως είναι μικρή ε, και είναι διαφορετική νομική οντότητα από τον όμιλο. Επίσης κύριε Επιτροπέ σωστό εσείς πολύ συχνά αναφέρεστε στην πρόληψη και βεβαίως η πρόληψη είναι καλύτερη αλλά και οπωσδήποτε πιο αποτελεσματική από την καταστολή αλλά αυτά τα πρόστιμα τα οποία γράφονται με μεγάλους τίτλους ε, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αποτελούν πρόληψη. Δεν νομίζω. Εάν αντί να αυξάνουμε τα πρόστιμα ε, αυξάναμε τον αριθμό των ελέγχων δεν θα είμαστε σε καλύτερο έδαφος πρόληψης. γιατί μερικές φορές στη Γαλλία τουλάχιστον τα πρόστιμα ε, είναι τόσο μεγάλα που χρειάζονται μερικές χιλιάδες χρόνια οι επιχειρήσεις έτσι ώστε να ξανασηκώσουν κεφάλι. Γι' αυτό λοιπόν ας μην βαυκαλιζόμαστε ε, με αυτά τα πρόστιμα. Ε, Βεβαίω η στρέβλωση του ανταγωνισμού και η παραποίηση των κανόνων του ανταγωνισμού δεν είναι ε, καλό πράγμα, αλλά βεβαίω και η επιβολή των προστήμων ε, θα πρέπει να είναι σωστή και τα πρόστιμα ε, θα πρέπει να είναι αντίστοιχα. Τώρα, μείωση των προστήμων, αν κατάλαβα καλά, είπατε όχι και είναι κρίμα. Ο κύριος Κίνερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν χρειάζονται κάτι αιώνες οι επιχειρήσεις για να πληρώσουν τα πρόστιμα, αλλά μου ακούγονται κάπως δρακόντιο αυτό το μετά. Κοιτάξτε, εγώ θα υποβάλω κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Αλμούνια για να μην ε, αυτοσχεδιάσω τώρα, αλλά θα ήθελα να φέρω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα πράγματι να κάνει η Κομισιόν μια αξιολόγηση αντικτύπου για τις καθητήριες γραμμές του 2006. Νομίζω μας είπατε πως κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω, ίσως πρέπει να με ενημερώσουν, αλλά θα χαιρόμουν να γίνει κάτι τέτοιο. Δεύτερον, ακούσαμε απόψε πως βεβαίως το βάρος δίνεται στα πρόστιμα. Πρόστιμα που επιβάλλονται σε εταιρείε παραβιάζουν τους όρους του ανταγωνισμού. Ναι, βεβαίω υπάρχει κλιμάκωση, αλλά δεν φαίνεται να του αποτρέπει αυτό. Εξακολουθούν να κάνουν τα ίδια. Πρέπει λοιπόν να είμαστε κάπω πιο εφευρετικοί στο τι κάνουμε. Όταν μιλάμε λοιπόν για τιμέ συνεννοημένε, συχνά μικρέ εταιρείε μπορεί να επηρεάζονται από τις μεγαλύτερες οι οποίες κάνουν ε, κάτι τέτοιο και χωρίς να φταίνε επηρεάζονται από αυτά τα πρόστιμα. Να σκεφτεί η Κομισιόν λίγο το κοινωνικό αντίκτυπο και ίσως θα μπορούσε να ευθύσει μια διαφορετική προσέγγιση στο Ηνωμένο Βασίλειο παραδείγματος χάρη επιτρέπει να μην μπορεί κάποιο πλέον να είναι διευθυντή, αντί να επιβάλλεται πρόστιμο στην εταιρεία. Έτσι δηλαδή ο υπέτειο πληρώνει μια έξυπνη προσέγγιση την οποία θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα είμαι σίγουρο, όπω ακούσαμε από άλλε χώρε. Εάν λοιπόν πάρουμε κάποιες πληροφορίε, θα μπορούσαμε έτσι να διασφαλίσουμε και τι θέσει εργασία στις εταιρείες εκείνες οι οποίες επηρεάζονται και αυτές από τι πρακτικέ των διευθυντών τους. Σας ευχαριστώ κύριε Σκίνερ. Η κυρία... Για ένα λεπτό κυρία Στήλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για αυτά που είπαν οι συνάδελφοι σήμερα εδώ. για τα πρόστιμα αυτά. Είναι για να σπάσουν τα καρτέλ που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και υπέρ του καταναλωτή. Αυτό που θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον Επίτροπο είναι το εξή, όπως είπε και ο κύριος Γκοζές και άλλοι. Θέλουμε πρόληψη πρώτα απ' όλα. Δεν πρέπει να δούμε στις διάφορες χώρες τι γίνεται. Η πρόταση του κύριου Σκίνερ όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Διευθυντή μια επιχείρηση. Μήπω είναι και αυτά πράγματα που πρέπει να δούμε εκτό από τα πρόστιμα, κύριε Επίτροπε. Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Στήλο. Ο κύριο ε, Κέλλη είναι ο τελευταίος, παίρνει το λόγο στο ΚΑΤΣΔΙ. Πολλά είναι τα άρθρα 101, 102 και 59 τα οποία ασχολούνται ε, με τον καθορισμό τιμών και βεβαίως ε, αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Ε, στο παρελθόν είχαμε μεγάλα προβλήματα Ας πούμε διαβάζω εδώ ότι ενώ ε, τα προστήματα 2009 αυξήθηκαν και παρά την, τις αποπληθωριστικές τάσεις ε, οι τιμές εξακολούθησαν να ανεβαίνουν. Ε, επομένως μόνο η κατανάλωση πέφτει, οι τιμές δεν πέφτουν. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε ξανά τις κατευθυντήριες γραμμές, να καθορίσουμε τάσεις σε μακρά χρονικά ε, διαστήματα και ε, μέσα σε αυτά τα μεγάλα χρονικά διαστήματα να καθορίσουμε τις κυρώσεις. Ο κύριος Σκίνερ έκανε, ε, καλή, έκανε μια καλή πρόταση, δηλαδή να πληρώνουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι, οι διευθυντές ας πούμε και τα πρόστιμα να είναι διαφοροποιημένα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο πάλι στον κύριο Μπανιέ, στον Επίτροπο, για την τελική απάντηση. Ευχαριστώ. Άκουσα τα επιχειρήματα και θα τα μεταφέρω στο συνάδελφο Χακίμ Αλμούνι. Μέσα από μένα και εκείνο δηλώνει ότι δεν πιστεύω ότι πρέπει σήμερα να προτείνουμε νέα νομοθεσία εντελώ καινούρια για τα πρόστιμα. Υπάρχει ο κανονισμός 1 του 2003 που σας είπα πριν και μπορεί να μας βοηθήσει για πολύ καιρό ακόμα. Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή τους και είναι ανοιχτή για κάθε πρόταση βελτίωσής τους. Οπότε αυτά τα οποία είπατε εδώ σήμερα είναι πολύ χρήσιμα. Κύριε Λένε, κύριε Γκοζές, κύριε Σκίνερ, δεν είμαστε κατά ελαστικότητας στους ελέγχους που κάνουμε για την εφαρμογή των κανόνων στα πλαίσια των καθηγητηρίων γραμμών και της νομολογίας, προκειμένου να λάβουμε υπόψη μας την δύσκολη οικονομική κατάσταση μερικές φορές. Πάντως όπως σας είπα και πριν ο κύριος Σαλμούνιο δεν βλέπει να υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών. Πιστεύει ότι οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές λειτουργούν καλά και έχουν αποδεχτεί αρκετά ελαστικές κατά τη διάρκεια της κρίσης. Μας επέτρεψαν να λάβουμε υπόψη μας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται ορισμένε επιχειρήσεις. Για τον υπολογισμό των προστήμων είμαστε δεσμευμένοι από τις διατάξεις που υπάρχουν και δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε χωρίς να έχουμε κάποια σοβαρή αιτιολογία. Αλλιώς τα δικαστήρια μπορούν να κυρώσουν την απόφασή μας. Κυρία Ταντεντβέλτ, άλλες λύσεις εκτός προστήμων πρέπει να δούμε σε τι βαθμό είναι εφικτό να τις ενσωματώσουμε στο σημερινό νομικό πλαίσιο αν είναι εναλλακτικέ ε, κυρώσει που υπάρχουν στα κράτη-μέλη, χρησιμοποιούνται από ό,τι ξέρω σε ελάχιστε περιπτώσεις και τα πρόστιμα είναι η κύρια κύρωση που υπάρχει. Αυτή η ιδέα υπάρχει. Ατομικές κυρώσει. έτσι κι δεν πρέπει να θέσουν σε αμφισβήτηση το σύστημα που έχουμε ελέγχου και τις επίκες. Επίσης, να εξετάσουμε το θέμα των μισθωτών των επιχειρήσεων και αν υπάρξει ατομική κύρωση δεν σημαίνει ότι συλλογικά η επιχείρηση δεν ε, πρέπει να υποβληθεί σε κυρώσεις εφόσον στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Πάντως οι σημερινοί κανόνες και η ομοιόμορφη εφαρμογή τους πιστεύουμε ότι είναι ένα μέσο αποτροπής τέτοιων μονοπωλιακών ε, συμπεριφορών μέσα στην ενιαία αγορά. Θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Έχουμε ένα διοικητικό σύστημα για να ε, φροντίζουμε να εφαρμόζονται καλά οι κανόνες ανταγωνισμού. Υπάρχουν πολλά πλέον εκτήματα. Υπάρχει νομολογία του δικαστηρίου που υποστηρίζει επίσης αυτό το σύστημα. Πριν αναφερθήκαμε και στην διαφάνεια. Ασφαλώς και ο συγητής και άλλη φορά τα έχουμε πει αυτά. Μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις. Είπαμε ότι οι καθετήριε γραμμές είναι ελαστικές. Και εξάλλου φέτος σας είπα ότι είχαμε και μια νέα πρακτική. των βέλτιστων πρακτικών. Κυρία Στήλερ και άλλοι αναφέρθηκαν ε, σε αναλεκτικές λύσεις. Μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά στα πλαίσια των ε, προγραμμάτων συμμόρφωσης. Εμείς πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις τα προγράμματα αυτά πρέπει να τα παίρνουν πολύ στα σοβαρά, κάτι το οποίο βοηθάει να αποφεύγονται παραβάσεις και έτσι στοιχίζει και λιγότερο το όλο θέμα. Τέλος, κύριε Σκίνερ και κύριε Κέλλη, αναφερθήκατε στις επιχειρήσεις που μερικές φορές υποφέρουν από τις κυρώσεις που τους επιβάλλονται και ότι δημιουργούνται και κοινωνικά ζητήματα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα διάφορα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό και προτείνουμε, όπως αναφέρεται και στη λευκή μας βίβλο, ότι επαληθεύουμε την αποτελεσματικότητα κάθε φορά που επιβάλλουμε κυρώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση για αυτό το θέμα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πίτρο Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτό το θέμα. Και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξη, που είναι οι παρεμβάσεις ενός λεπτού. Έχουν ζητήσει διάφοροι το λόγο για να